Χαίρετε. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα σας πρότεινα να αρχίσουμε από το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, γιατί απουσιάζει η κυρία Κρίστα Ρόβολ. Α, παρευρίσκεται. Μα γιατί με παραπληροφορείτε πάντα. Liebe, Έχεις μια στιγμή να, καιρό να μείνεις να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Πρέντα. Γιατί κανονικά θα πρέπει να αποχωρήσει νωρίτερα και μετά ε, να αλλάξουμε με το δικό σου θέμα. Εντάξει. Και ερχόμαστε λοιπόν στην έκθεση πρόοδου για την Ισλανδία για το 2011. Ο εισηγητή μα, ο κύριο Κρίστιαν Τραν Πρέντα, θα μα κάνει την εισαγωγή. Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον που έδειξαν κατά τη διάρκεια της πρώτης συζήτησης που είχαμε για την Ισλανδία Και φυσικά για το ενδιαφέρον που έδειξαν υποβάλλοντας τόσες ε, τροπολογίες, 62 στο σύνολο. Εγώ πρότεινα πέντε συμβιβαστικές τροπολογίες. Μία συμβιβαστική ξεκινώντας με την παράγραφο 4 για τη συνταγματική μεταρρύθμιση που γίνεται στην Ισλανδία. Δεύτερη συμβιβαστική για την παράγραφο 9 του αρχικού ψηφίσματος. για τον πολιτικό διχασμό που βλέπουμε εντό της ε, κυβέρνησης αλλά και μεταξύ των κυρίων ε, πολιτικών κομμάτων της Ισλανδίας γιατί εντός της κυβέρνησης υπάρχει αντίθεση, αλλά και εντός των κυρίων των μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων. Έπειτα, η τρίτη συμβιβαστική, παράγραφος 12, σχέσεις της Ισλανδίας με την Ένωση μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τέταρτη συμβιβαστική αφορά την παράγραφο 13 και αναφέρεται σε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υιοθετήσει η Ισλανδία έτσι ώστε να πληρεί τα κριτήρια ένταξης και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την άρση του προστατευτισμού σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Και τέλος, η πέμπτη συμβιβαστική αφορά την παράγραφο 20. Και έχει να κάνει με την ε, σημερινή φάση της Ισλανδίας στην ενταξιακή διαδικασία και πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις ανάγκες πλήρωσης ε, εξέτασης διαφόρων κεφαλαίων μέσα στην πορεία της ε, ένταξης. Οι υπόλοιπε τροπολογίε, ε, οι περισσότερε υποστηρίζουν το κείμενο και το διευκρινίζουν. Δεν μπορώ όμω να, να δεχτώ τι τροπολογίε του κ. Μάντελον που θέλει να θέσει τέλο στι διαπραγματεύσει. Γιατί σε αυτή τη φάση στην Ισλανδία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και εμεί την ίδια ιδέα. Τη συνέχιση του δηλαδή και μάλιστα καθώς η σημερινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ολοκληρώσει την εξέταση των διαφόρων κεφαλαίων μέχρι τα τέλη της Δανικής Προεδρίας της Ένωσης. Περιμένουμε μέγα ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις και τις αντιδράσεις των συναδέλφων. Εγώ υποστηρίζω τον διορισμό ενός νέου σκεώδου συζητητή από την ε, Μάρα των Σοσιαλιστών, τον συνάδελφο και φίλο κύριο Παντζέρη. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Εγώ αντικαθιστώ τον κύριο Σασόλη που ανέλαβε άλλες, άλλα καθήκοντα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέντα για την πολύ ισορροπημένη έκθεση που μας παρουσίασε και επειδή συμπεριέλαβε στις συμβιβαστικέ τροπολογίες την θέση της ομάδας των σοσιαλιστών δημοκρατών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των τομέων που δεν καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Και έπειτα ε, την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών ανάμεσα στην Ισλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΕΟΧ καθώς και την ευχή ότι οι διαπραγματεύσεις οι προενταξιακές θα συνεχίσουν με ικανοποιητικό τρόπο κατά τη διάρκεια και θα ολοκληρωθούν στη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Ο κύριος Πρέντα έκανε εξαιρετική δουλειά και νομίζω πως μπορούμε να συνεργαστούμε για να ορίσουμε όσο γίνεται πιο ε, ομόφωνη θέση καταρχήν στην Επιτροπή μας και έπειτα στο σύνολο του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Κανεί άλλο δεν θέλει το λόγο. Έχω μια ερώτηση στον άλφο Πανσέρη, γιατί πριν από λίγε μέρε ήρθαν στο γραφείο μου εκπρόσωποι ε, του ναι ε, στο δημοψήφισμα μπορεί να ε, είναι η πλειοψηφία του λαού υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων, αλλά υπέρ της ένταξης φάνηκε ότι είναι μόνο το 37%. Ε, τι ενδείξει έχετε ότι θα γίνει πλειοψηφία και ποια είναι τα προβλήματα βασικά, τα θέματα της αλίας και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τι μπορεί να γίνει για να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό πλαίσιο. Γιατί θα ήταν δυσάρεστο. Μετά από δύο φορές διαπραγματεύσεις είχαμε ε, στην Ορβηγία και τελικά δεχτήκαμε απόρριψη. Τώρα μην πάθουμε τα ίδια και με την Ισλανδία. Θα με ενδιέφερε λοιπόν η δική σας ε, εκτίμηση, ο εισηγητής. Ε, Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια σας, ε, κύριε Παντζέρη, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. οι αντιρρήσεις για την προσχώρηση της Ισλανδίας βασίζονται σε διάφορα αίτια ιστορικά. Από μια, μια κάποια αίσθηση αυτάρκειας και η θελημένη απομόνωση από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά Υπάρχει και ένας λόγος που δεν ε, προέρχεται από την ιστορία, αλλά από του σύγχρονους καιρού. Το βασικό επιχείρημα υπέρ της ένταξης της Ισλανδίας είναι ότι μάλλον υπέρ της ένταξης, ναι, ήταν η αδυναμία του Ισλανδικού νομίσματος, της Ισλανδικής κορώνας, απέναντι στο ευρώ. Όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, το κύριο επιχείρημα των υποστηρικτών της ένταξης ήταν η ισχύς του ευρώ απέναντι στο Ισλανδικό νόμισμα. Ενώ τους τελευταίους μήνες, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη, το επιχείρημα αυτό και οι ισχύς του έχουν αποδυναμωθεί. Για την ώρα δεν έχει προβληθεί κάποιο άλλο αντίστοιχο επιχείρημα στην κοινή γνώμη της Ισλανδίας. Δηλαδή, από τη μια πλευρά έχουμε αυτούς τους παλιούς ιστορικούς λόγους, ε, για ότι η Ισλανδία δηλαδή μπορεί να είναι αυτάρκης και είναι ικανοποιημένη με αυτά που έχει, με τη συμμετοχή της δηλαδή στον ΕΟΧΟ και στο Σέγγεν και μπορεί να διατηρήσει την ε, απόλυτη κυριαρχία της. Ε, και από την άλλη, έχουμε ένα επιχείρημα το οποίο αποδυναμώθηκε με τα όσα συμβαίνουν στην Ένωση. Αυτό το επιχείρημα δηλαδή που έλεγε ότι το βασικό πλεονέκτημα της Ισλανδίας θα ήταν το ευρώ από την ε, ένταξη. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς? Α, ναι. Πρόεδρε, ο συνάδελφο Παντζένη, ο σκιώτη ε, για την ομάδα μα. Παντσέρι. Παντσέρι. Και ο σκιώτη ε, από την ομάδα μα. Νομίζω ότι μας ανέφερε τι ε, απόψεις μας για τη συμφωνία αυτή, αλλά θα ήθελα να μας ενημερώσετε για τη συζήτηση που διεξάγεται στην ε, Ισλανδία για τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και αν θεωρούν ότι η προσχώρηση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τη χώρα. Η κυρία Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή Κρίστιαν Πρέντα για την ε, πολύ καλή αυτή έκθεση που είναι πολύ ισορροπημένη. Συμμετείχα στην ε, σχετική αντιπροσωπεία που επισκέφτηκε την Ισλανδία την προηγούμενο έτος, τον Οκτώβριο αν δεν κάνω λάθος. Και ήταν σαφές ότι στο εσωτερικό της χώρας ε, μόνο μία συμμαχία σοσιαλδημοκρατίας είναι υπέρ της προσχώρησης της Ισλανδίας της Ένωσης όλα τα υπόλοιπα κόμματα, οι πράσινοι και η ανεξάρτητοι, η προοδευτικοί, το κόμμα της κίνησης που όλοι συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική αντιπολίτευση αντιμετωπίζουν το διχασμό σε ό,τι αφορά την προσχώρηση στην Ένωση. Κάποιοι από την αντιπολίτευση λοιπόν ε, θεωρούν και μας το εξέφρασαν τότε ότι θα πρέπει η Ισλανδία να αποσύρει την αίτησή της για την προσχώρηση στην Ένωση. Θεωρώ ότι με τις διαπραγματεύσεις ε, τις αξιακές ως μέσο η αντιπολίτευση αποδυναμώνει την θέση της Ισλανδίας στις διαπραγματεύσεις ε, απειλώντας να φύγει από το Κοινοβούλιο, απειλώντας με Και γι' αυτό λοιπόν πρότεινα τις τροπολογίες αυτές και νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειώσουμε αυτή την μετακίνηση της Ισλανδικής ε, κυβέρνησης. Ε, η αλλαγή μάλλον ο σχηματισμός της ε, Ισλανδικής κυβέρνησης μας δίνει κάποιες ελπίδες για πιο μεγάλη δέσμευση σε ό,τι αφορά την πρωταξιακή και την ενταξιακή διαπραγματε... διαπραγματεύσεις. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι το εξή. Όπω ξέρουμε, οι πληροφορίε είναι σημαντικέ, κρίσιμε. Καλωσορίζω λοιπόν την ε, εκκίνηση, την έναρξη του σχετικού γραφείου πληροφόρηση στην Ισλανδία που θα δώσει στους πολίτες στην Ισλανδία όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με το τι σημαίνει η ένταξη τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ισλανδία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ρητά τον εισηγητή για την τόσο επικοδομητική στάση που επέλεξε για την έκθεση αυτή και πραγματικά αντικατοπτρίζει το επικοδομητικό πνεύμα που πριτάνευσε και στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Ισλανδίας ε, γενικά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με την τροπολογία και ε, αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι εξή πτυχή. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων βεβαίως θα κληθεί ο λαός της Ισλανδίας ανεπηρέαστος από οποιαδήποτε θέση, ε, οποιοδήποτε σχηματισμού να ψηφίσει σε δημοψήφισμα και να μην επηρεάζεται ούτε από το ναι ούτε από το όχι. δεν ξέρω κατά πόσο είναι σκόπιμο να υποστηρίζουμε τη μία ή την άλλη άποψη, το ναι ή το όχι. Θα πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος, γιατί έτσι θα εκφράσουν και τα βαθιά τους ε, δημοκρατικά αισθήματα που μπορεί να είναι ε, τελικά προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να βγάλει τα συμπεράσματά της και για μελλοντικές ε, διευρύνσεις και για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης. Ο κύριος Φαν Μπάλεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για το έργο του που θα μας βοηθήσει όλους εμάς τους κοιόδες. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Περιλαμβάνεται άλλωστε και στις τροπολογίε. Αλλά για την Ισλανδία θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι οι υποχρεώσει ε, που εμπλέκονται στην περίπτωση τη ε, τράπεζα ISAVES εξακολουθούν να υφίστανται. Άρα τι σημαίνει αυτό ότι για να προσχωρήσουν την Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσουν και να ε, συμμορφωθούν με την απόφαση του δικαστηρίου της ΕΦΤΑ που είναι ανεξάρτητο δικαστήριο. Δες, Ο κύριος Πρέντα. Uh, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους και για τις ερωτήσεις που έθεσαν. Σύντομα, να πω για την ερώτηση της κυρίας Γκόμες. Πρέπει να σας πω ότι στην Ισλανδία η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της Αρκτικής θεωρείται θετική, η εμπλοκή μάλλον της Ένωσης. Και γιατί, γιατί σε αυτή τη φάση η Ρωσία, η ΙΠΑ και η Νορβηγία προσπαθούν να προβούν σε αποφάσεις αγνοώντας την Ισλανδία, αγνοώντας τη μικρή αυτή χώρα. Όμως η πολυμερής μας ε, θέση εκλαμβάνεται θετικά από τον Ισλανδικό λαό και θεωρούν πως έτσι βρίσκονται σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι μέσα στους ε, ε, αντίθετους στην προσχώρηση επικρατεί η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει την Ισλανδία μόνο και μόνο για να ευνοήσει την θέση της ως προς την Αρκτική. Ορισμένοι μάλιστα θεωρούν ότι έχουμε απλά κάποιο κρυφό σχέδιο για να, καλύψουμε, για να έχουμε μάλλον καλύτερη θέση στον διάλογο περιεκτικής. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της κυρίας Αντρική Ενέν, οι αλλαγές που γίνονται εντός της κυβέρνησης δεν έχουν μεταβάλει τι ε, αρχέ περί συνέχιση ε, των διαπραγματεύσεων. Είναι αλήθεια ότι οι αλλαγέ κατά τη διάρκεια αυτού του ανασχηματισμού στο επίπεδο του, Υπουργείου, του Υπουργικού Συμβουλίου οι αντίθετοι στην προσχώρηση έχουν έναν λιγότερο στην κυβέρνηση. Ο κύριος Γιάννεσεν αποσύρθηκε από την κυβέρνηση. Ήταν ένας από τους πιο ε, κραυγαλαίους αντίπαλους της προσχώρησης, της ένταξης. Πιστεύω λοιπόν πως αυτό είναι ένα μήνυμα για, από πλευρά τη κυβέρνηση ότι δηλαδή η εμπλοκή στι διαπραγματεύσει θα είναι πιο συνεπή πλέον. Για τι παρατηρήσει του κυρίου Σόλτ, θα ήθελα καταρχήν να σα θυμίσω το γεγονό ότι όταν η Ισλανδία αποφάσισε να ζητήσει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσισε ότι στο τέλος, αποφασίστηκε μάλλον στο τέλος των διαπραγματεύσεων θα γινόταν δημοψήφισμα. Αυτό έχει ήδη λοιπόν αποφασιστεί. Και αν τα πράγματα πάνε καλά, στα τέλη αυτής της διαδικασίας θα γίνει ένα δημοψήφισμα όπου ο Ισλανδικός λαός θα έχει λόγο. Όσον αφορά τη συζήτηση για την Ισλανδία, πιστεύω πως ε, σε αυτή τη φάση η ευρωπαϊκή στάση είναι αμερόληπτη. Εμείς ακούμε τα υπέρ και τα κατά αλλά οι αντίπαλοι της ένταξης είναι περισσότερο παρόντες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από ότι υποστηριχτές της ένταξης για λόγους που οφείλονται στην ιστορία της χώρας. Τέλος, για τις παρατηρήσεις του κυρίου Φαν Μπάλεν για το iSafe. Να θυμίσω ότι η Ισλανδική κυβέρνηση έχει ήδη πληρώσει το 1 τρίτο του χρέους που είχε προς τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και των, ε, των, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου με και των κάτω χωρών. Και όσον αφορά την απόφαση του δικαστήριου της ΕΖΕΣ, υπάρχει συνένεση στην Ισλανδία και η κυβέρνηση στηρίζει τα όσα ανέφερε ο κ. Φαν Μπάλεν. Ε, θα ήθελα ωστόσο να κλείσω αυτή τη συζήτηση πριν να σας καλέσω στην στα εγγένεια της έκθεσης την οποία φιλοξενώ εγώ στο κτίριο εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για την ε, υπέροχη Ισλανδία. Για τα εγγένεια αυτά θα γίνουν αύριο το απόγευμα στις 6.30. Είναι ακόμα ένας τρόπος για να γνωρίσουμε καλύτερα την Ισλανδία που είναι υποψήφια χώρα που όπως γνωρίζετε προσπαθεί να ε, κλείσει τα κεφάλαια μέχρι τα τέλη της Δανέζικης Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας και τις υπόλοιπες τροπολογίες. Θα τις συζητήσουμε στην έκθεση εκεί που θα έρθουμε να δούμε. Επανερχόμαστε στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης και θα Παρακαλούσα την κυρία Κρίστα Τρόβολ να μας κάνει την εισαγωγή για το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής εμπορική και επενδυτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μεσογειακό Νότο μετά την Αραβική Άνοιξη. γνωμοδότηση είναι ε, αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου που συμμετέχει η κυρία Κουίσταουτ επίσης και είναι δεδομένη η συνέχεια και η ολότητα και η πληρότητα της έκθεσης. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η Αραβική Άνοιξη αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την επικοδομητική μας δέσμευση στις χώρες της Αραβικής αυτής επανάστασης ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολιτική ευθύνη και αυτό θα πρέπει να περάσει και στις πράξεις, να μην μείνει στα λόγια. Άρα, η Επιτροπή Εμπορίου προετοίμασε μία έκθεση πρωτοβουλία στο εμπόριο για την αλλαγή, υπέρ της αλλαγής και έτσι υποστηρίζει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση του εμπορίου με τις χώρες αυτές. Το πρώτο θέμα αυτό, ε, στο πρώτο θέμα μάλλον στο πλαίσιο αυτό, θα είναι να βελτιώσει το κλίμα για τις επενδύσεις. Γι' αυτό λοιπόν σας παρουσιάζω την σχετική γνωμοδότηση για την Επιτροπή Εμπορίου τονίζουμε και υποστηρίζουμε τις βασικές δημοκρατικές αρχές στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Μιλάμε για την ελευθερία θρησκείας, ε, πίστης, συνείδησης. Πρόκειται για τις ε, πλέον καθολικές ε, αξίες, θεωρώ, αλλά υποστηρίζουμε και καλούμε τη μεταβατική κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν να περάσει σε μια ειρηνική δημοκρατική κατάσταση. Καλούμε και τις κρατικές αρχές των μεμονωμένων κρατών να σέβονται τα δικαιώματα του λαού για ειρηνικές διαδηλώσεις και να να καταδικάζουν οποιαδήποτε είδη καταστολής. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε την σημασία των ελεύθερων εκλογών για την διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Η πολιτική σταθερότητα, ωστόσο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, αλλά η πολιτική σταθερότητα ενισχύεται μέσω της οικονομικής ευημερίας, μέσω της ανάπτυξης στις περιοχές αυτές. Αναλόγως λοιπόν και αντίστοιχα, θεωρώ ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τους όρους εκείνους με τους οποίους μπορούμε να επενδύσουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Και για να πετύχουμε το στόχο αυτό υπάρχουν κάποια πρώτα μέτρα και κάποιες πρωτοβουλίες, όπως κάποια προγράμματα τα οποία ήδη υφίστανται. Αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν και να επεκταθούν, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και καλός συντονισμός. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εκείνους που υπέβαλαν τροπολογίες οι οποίες υποδεικνύουν ακριβώς αυτή την ανάγκη και την υποχρέωση συντονισμού των πρωτοβολιών. Υπάρχει και μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΠΑ της ε, εκπροσώπου για μια, με τίτλο ε, μια νέα αντίδραση σε μια γειτονιά που αλλάζει». Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να τονίσουμε πώς ε, κάποιες τέτοιες αρχές θα πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη. και την πρωτοβουλία ε, της ε, Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκή Ένωση την Ισία για την καλύτερο συντονισμό της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Υποστήριξης της ε, χώρας. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επενδυτή. Γιατί στην παρούσα φάση συζητάμε θέματα μετάβασης σε ό,τι αφορά την προστασία των άμεσων επενδύσεων και τη μεταφορά τους από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό θα αποτελούσε ένα τομέα εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι αφορά την επέκταση, την διεύρυνση μάλλον των ε, ε χρηματοοικονομικών σχέσεων με τους ε, γείτονες προς τον Νότο. Ε, κατατέθηκαν 67, ε, 17 τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και θα κάνω κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Ελπίζω να βρει σύμφωνος τους ε, ε, συναδέλφους και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρωθεί το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Εγώ σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφε. Μια σειρά συνάδελφων έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Ρομέρο πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε ζήτησα το λόγο για την έκθεση αυτή, που είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας, διότι για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική αυτή η έκθεση και να δημιουργηθεί πραγματικά ένας χώρος ελευθέρων συναλλαγών στη Μεσόγειο. Και θυμίζω ότι ήταν και το όνειρο της διάσκεψης της Βαρκελόνης το 2010 ήδη η ε, Μεσόγειος να ήταν χώρος ελευθέρων συναλλαγών. Ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αυτό το όνειρο. Είναι προφανές ότι οι επαναστάσεις στον αραβικό κόσμο δημιούργησαν νέα δεδομένα και οι σχέσεις μας πρέπει να είναι διαφορετικές πλέον. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται μελέτη σκοπιμότητας και αντικτύπου. Δηλαδή, οι χώρες αυτές που είναι στο νότο της Ευρώπης και παράγουν γεωργικά προϊόντα, τα προϊόντα τους θα έχουν επιπτώσεις ε, στις νότιοευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχη παραγωγή. Εγώ είμαι από την Ανδαλουσία και ε, στην περιοχή μου γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις και διαμαρτύρονται οι πολίτες για τη συμφωνία που είχαμε για γεωργικά προϊόντα. Τα ίδια μπορούν να συμβούν στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Νότια Γαλλία, διότι πραγματικά τα προϊόντα του Νότου είναι πιο ανταγωνιστικά, είναι πιο πρόημα των χωρών της Νότιας Όχθης Μεσογείου και θα πρέπει να γίνει μελέτη αντικτύπου πώς θα επηρεαστεί η γεωργική παραγωγή των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Αυτό το θέμα δεν είναι καινούριο. Όταν θέλησε να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή κοινότητα η Ισπανία, μας απέριπτε η Γαλλία και είχαμε πολύ μακρά μεταβατική περίοδο. Και χρειάστηκε να την ολοκληρώσουμε και ακόμα και έτσι οι Γάλλοι πετούσαν τα φορτηγά με τις ντομάτες, τα βιάζαν στους δρόμους και ό,τι θέλαμε εμείς να εισάγουμε στην Ευρώπη ε, και να εξάγουμε από την Ισπανία. Έχει συμβεί αυτό λοιπόν, έγιναν διαδηλώσεις ε, για τη γεωργία, αλλά στο μέλλον μπορούμε να το δούμε και σε άλλους τομείς, ε, το τομέα της παραγωγής τροφίμων και άλλων. Χρειάζεται λοιπόν μελέτη αντικτύπου να δούμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε να είναι ε, συμπροματική αυτή η παραγωγή και η εισαγωγή. Ωραία είναι να τα λέμε, αλλά εκείνοι που έχουν παραδοσιακή γεωργία δεν έχουν καταλάβει την ιδέα. Παρόλο που επενδύουν δικοί μας επενδυτές από το νότο της Ευρώπης στο νότο της Μεσογείου, χρειάζεται μεταβατική περίοδος μακρά που θα έχει και πολλά αρνητικά αποτελέσματα στη φιλοευρωπαϊκή στάση και αισθήματα των λαών του Νότου. Και θυμηθείτε, η ευρωπαϊκή ε, κοινότητα γεννήθηκε για να προστατεύσει τους αγρότες μετά την ΕΚΑΧ βεβαίως. Είναι η πιο ευάλωτη τομή και θα πρέπει, όσο και είναι έκθεση πρωτοβουλίας, να έχουμε υπόψη μας το γεγονός ότι αυτό μπορεί να ε, εμφανιστεί και ο δρόμος να είναι πάρα πολύ μακρύς. Τελεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σάκε. Uh, Ευχαριστώ. Εγώ παίρνω σύντομα το λόγο γιατί ο σκιώδης ε, συγγετής ο ε, κύριος Σάρνες, δεν είναι εδώ. Αλλά πιστεύω πως η συνεργασία με τον συγγετρία ήταν ε, επικοδομητική και καρποφόρα και μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Θέλουμε μόνο να ρωτήσουμε αν μπορούμε να προσθέσουμε στη συμβιβαστική τρία ότι ο κύριος Σάρνες υπογραμμίζει ότι υπάρχει, ότι είναι σημαντικό να συνεργάζονται τα επενδυτικά σώματα, όπως υπάρχει και στην τροπολογία 12. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω, εκτός αν θέλετε, αλλά αυτές είναι μόνο οι παρατηρήσεις του κυρίου Σαρνέζ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάιρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κουίσχαουτ για την γνωμοδότησή της. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό που ζητεί από τις εθνικές αρχές να σέβονται το δικαίωμα των λαών να διαδηλώνουν ειρηνικά και να μην ε, προχωρεί σε βία η καταστολή. Επίσης ε, ζητά ανοχή, σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ελευθερία της έκφρασης, ανεξιτρισκεία. Επίσης η νέα μεμονωμένη ετομική εστίαση είναι σημαντική, το εξήγηλε και η κυρία Άστον για μια νέα γειτονία και επίσης την ανάγκη να μειωθούν οι ανισότητες και οι κοινωνικές και οι εδαφικές. Κάτι που λείπει όμως, δεν δίνεται αρκετή έμφαση στα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα που έχει μεγάλη σχέση με τα όσα είπε η κυρία Ρομέρο. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε υψηλές απαιτήσει για κοινωνικά δικαιώματα, για ιχνηλασιμότητα. Όλα αυτά δεν υπάρχουν στις χώρες της Νότιας Όχθης Μεσογείου και είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Θα πρέπει αυτά τα κοινωνικά δικαιώματα να επιβαρύνουν εξίσου τους παραγωγούς εκεί και τους ε, κατασκευαστές ε, προϊόντων, που δεν είναι βάρος, είναι δικαίωμα για τους εργαζομένους. Επίσης, κάτι άλλο μου λείπει που ζήσαμε ως εμπειρία και στην Αραβική Επανάσταση. Το άρθρο 2 ε, τη συμφωνία σύνδεση και να συνδέεται με αυτού του όρου. Δηλαδή θα πρέπει να διδαχθούμε από τα σπάλματά μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διατήρησε ακέραιες ε, τι συμφωνίε σύνδεση με τα καθεστώτα Μπέναλή και Μουμπάρακ και θα πρέπει να διδαχθούμε σε τέτοιε καταστάσει, τέτοιες εμβέλειες θα πρέπει να υπάρχει αιρεσιμότητα και να είναι αμοιβαία εγγύηση για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ πολύ.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 είναι καλό το σχέδιο έκθεση, αλλά υπάρχουν δύο σημεία που νομίζω θα πρέπει να υπογραμμιστούν κάπω περισσότερο και να ευαθυνθούν. Καταρχήν, αυτό που κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να καλέσουμε εντόνω όλε αυτέ τι χώρε σε μια διαδικασία περιφερειακή ολοκλήρωση, διότι αυτή είναι μια ουσιαστική προπόθεση για να υπάρξει δυνατότητα ανάπτυξης ε, τη οικονομία, του εμπορίου, τη κοινωνία και των υποδομών. Δεύτερο θέμα, επί τη των όσων έλεγε και η Κάρμεν Ρομέρο, ίσως ε, μέσω της ανάγκης εντοπισμού ε, θεμάτων ε, εμβάθυνσης για τη διαδικασία ελεύθερων συναλλαγών και στον αντίκτυπο που θα έχει αυτό για το σύνολο των μεσογειακών χωρών. Αυτή η εμβάθυνση είναι σημαντική για να είναι θετικές οι επιπτώσεις, ο απόίχο και να ικανοποιήσουν, να ωφελήσουν όλους. Ευχαριστώ. Lucky. Σαρλάκη. Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής της ε, ομάδας και ε, των σοσιαλιστών και υποστηρίζουμε αυτή την ε, γνωμοδότηση θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω κάτι που ήδη έχει ε, τονιστεί, ότι υπάρχει γενικά μεγάλη καθυστέρηση από πλευρά της Ένωσης όσον αφορά μια αξιόπιστη στρατηγική για τις χώρες που έζησαν αυτήν την αποκαλούμενη Αραβική Άνοιξη. Μετά από ένα χρόνο δεν έχουμε τίποτα περισσότερο παρά κάποιες αόριστες ιδέες, λόγια δηλαδή, που και, και ελάχιστες απαντήσεις σε πολύ πιεστικά και συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι θέματα τα οποία ήδη τόνισαν οι συνάδελφοι. Τι είδου ανάπτυξη θέλουμε να ευνοήσουμε σε αυτές τις χώρες. πώ θα λύσουμε το ζήτημα του ανταγωνισμού με τις νότιε ευρωπαϊκές παραγωγές. Τι είδου γεωργία θέλουμε να γίνει. Τι είδου ε, αλλιευτική βιομηχανία, αν μείνει καμία, ε, θα στηρίξουμε αν λάβουμε υπόψη την τεράστια προμήθεια, παροχή μάλλον Ε, αλλιευμάτων και τον μεγάλο αλλιευτικό στόλο σε ολόκληρη την Μεσόγειο. Πώς θα αποφύγουμε τον ανταγωνισμό με αυτές τις χώρες από τη στιγμή που θα αρχίσουν να, να πορεύονται σε ένα αξιόπιστο ε, μονοπάτι ανάπτυξης. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα θα παραμένουμε στην συνηθισμένη θέση κάποιου που έχει πολύ καλές προθέσεις αλλά δεν είναι αξιόπιστος και δεν έχει συγκεκριμένες ιδέες να υπογραφεί. Ένα χρόνο μετά την Αραβική Άνοιξη εξακολουθούμε να καλούμε, να προσκαλούμε, να αναπτύξει, λέει, η Κομισιόν στρατηγικές για επενδύσεις κτλ. Πολύ ωραία όλα αυτά στα λόγια, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι και πιο πιστικοί στα τι θέλουμε να κάνουμε. Πριν από έξι μήνες ένα σωρό ιδέες ακούστηκαν για το πώς θα κινητοποιηθούν πόροι, κάναμε λόγο για ένα σχέδιο Marshall για τη Βόρεια Αφρική και την ε, Μέση Ανατολή, για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των πρώην τυράννων ε, για, ως πόρο για την ανάπτυξη, αλλά τελικά ελάχιστη συνέχεια έχει δοθεί ε, σε όλα αυτά τα συγκεκριμένα, ιδέες και μάλιστα κάποιες φορές φοβούμε πως επανερχόμαστε στην αφετηρία και ωστόσο υποστηρίζω αυτή την ε, έκθεση. Έχουμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες ε, σε όχι θεμελιώδη ζητήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γκράισλερ Ντόφλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ ειλικρινά ε, την εισηγήτρια. Θα πρέπει οπωσδήποτε, και είναι κατεπήγον αυτό, τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη αυτά. Ε, οι επαναστατικές διαδικασίες έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Μόνο μετά την ολοκλήρωσή τους γνωρίζουμε πώς θα μπορέσει να προχωρήσει μια χώρα. Αν είδα τι έγινε ε, στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση, τα κράτη είναι μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ε, σύμμαχοί τους, ε, από την Πολωνία μέχρι τη Βουλγαρία αγωνίζονται και παλεύουν ακόμα 22 χρόνια. Τραβάει λοιπόν σε μάκρος αυτό και σε βάθος. Καλό είναι να θέλετε μελέτη αντικτύπου, αλλά εάν δεν αντιδράσουμε και δράσουμε γρήγορα, τότε δεν θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τις συνέπειες. Μιλάμε για τη γεωργία. Εγώ είμαι 17,5 ε, χρόνια εδώ βουλευτής και βλέπω ότι γίνεται. Από το Σίκο Μάνσχολτ από τη δεκαετία του 60 και του 70 για τη γεωργία συζητάμε και ασχολούμαστε. Ε, με το Φίσλερ ε, βελτιώθηκε η κατάσταση. Ήταν η μεταρρύθμιση του Μαξάρη και του Μάνσχολτ πραγματική καταστροφή. Κοιτάξτε τις μονοκαλλιέργειες από τη Σεβίλη και πέρα όλες τις ελιές ε, και πώς έχει καταστραφεί η κατάσταση. Με πιάνουν τα κλάματα. Ε, όταν πας με αεροπλάνο στην Αδαλουσία δεν βλέπεις τίποτα παρά μόνο ε, τους μουσαμάδες από τα ε, θερμοκήπια. Αυτό δεν είναι γεωργία. Θα ήθελα πραγματικά εγώ να εισηγηθώ να αναπτυχθεί και ο κρατικός τομέας στις χώρες αυτές για να μπορέσουν να θρέψουν τον πληθυσμό τους. Κάντε λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε πώς θα διαρθρώσουμε τις δικές μας εξαγωγές και να τους αγοράζουμε και προϊόντα, γιατί θα πρέπει ε, για να αναπτυχθεί μια χώρα να δημιουργεί εισόδημα για να καλύπτει και τις άλλες ανάγκες και τις τεχνολογικές. Έχετε πάει στην Αίγυπτο. Εγώ πήγα πριν από δύο χρόνια και γνωρίζω και τις άλλες χώρες. Είναι πάρα πολύ εκρηκτική η κατάσταση και ολέθρια της φτωχής ε, ε κοινότητα. Άμα πάτε στο Κάιρο μην πάτε μόνο στα μουσεία και στις πυραμίδες και κουνάτε σημαίακια στην πλατεία Ταχρήρ. Πηγαίνετε λίγο και στις φτωχογειτονιές να δείτε τι γίνεται. Και στην πολιτική αλληλεία στο κάνουμε αυτό. Ελπίζω να βοηθήσουμε, αλλά να συζητήσουμε και για την ανοιχτή μετανάστευση, να μπορούν να έρχονται οι άνθρωποι. Έχουμε τεράστια προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας μην γελιόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κατεβάσουμε τα ρολάκια να πούμε τέρμα επειδή έχουμε εμεί προβλήματα. Θα τα βρούμε μπροστά μας, θα μεταφερθούν και τότε θα σπάσουμε πλάκα, για να το πω έτσι, ομά. Θα πρέπει πραγματικά να κινητοποιηθούμε γιατί δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε και το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ε, κυρία Γκόμα, σας ευχαριστώ για τις καλές σκέψεις που εκφράσατε. Uh, uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε αρκετοί συνάδελφοι από την ομάδα μας και ο Σκιωδής μας υπέτυξαν πολλά σημαντικά στοιχεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Θα ήθελα να τονίσω επίσης αυτά που ακούσαμε, ότι δηλαδή θα πρέπει η Επιτροπή μας και το Κοινοβουλίο μας να ζητήσει μια εις ε, μελέτη για τον αντίκτυπο όχι μόνο στο θέμα της γεωργίας, της βιομηχανίας, της αλληλείας, αλλά και σε άλλους τομείς με μεγάλο δυναμικό. Μεγάλο δυναμικό και θετικό ως προς το όφελος, αλλά και ε, δυναμικό σύγκρουσης. Και έχω υπόψη με τον τουρισμό και την ενέργεια. Η ενέργεια όχι μόνο το αέριο και το ηλεκτρικό, αλλά και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν πολλά Υπάρχει μεγάλο δυναμικό και σε ό,τι αφορά τη σύνδεση ενδεχομένω ε, τη Βόρεια Αφρική με την Ευρώπη, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν από μια σχετική τέτοια μελέτη. Και θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Θα έπρεπε και η Επιτροπή μας να τονίσει αυτές τις πτυχές. Επίσης, η αρχή του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον επενδυτικό για την ανάπτυξη των επενδυτικών σχέσεων χωρίς κράτος δικαίου. Και πάλι νομίζω ότι θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Καταλαβαίνω πώς αναφέρει ο εισηγητής την ανάγκη να υπάρχει μικρότερο σχέδιο, αν θέλετε. Αλλά θα θέλαμε και πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι το σημαντικό είναι να υποδείξουμε προς την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ότι θα την πάρουμε στα σοβαρά και ότι θα αξιολογήσουμε ανα πάσα στιγμή κατά πόσον τα σχέδια αυτά εφαρμόζονται. Νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο ίσως στην παρούσα φάση να μας δώσουν πιο πολλέ λεπτομέρειες. Τέλος, να τονίσω τη σημασία του να αναφερθεί κάπου η συμμετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, στο παραγωγικό δυναμικό. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό, αν θέλετε, τεστ για το κατά πόσο οι γειτονικέ αυτές χώρες μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το ταλέντο που πολλές φορές πάει χαμένο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όπως ξέρετε στις πιο πολλές από αυτές τις κοινωνίες η συμμετοχή των γυναικών, η πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και δημοκρατική ζωή θα αποτελέσει το κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο θα υπάρχει πραγματική δημοκρατική μετάβαση ή όχι. Ο κύριος Μιγιάν Μον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια για το κείμενό της και για την προθυμία της ε, να συμπεριλάβει τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Είναι λίγες, ε, αν θυμάμαι, από τις 17, οι δικές μου είναι τέσσερις και από τις ε, συνομιλίες που είχα μαζί της και το email που μου έστειλε κατάλαβα ότι θα τις λάβει υπόψη της και στους συμβιβασμού για την καλοσύνη. Θέλω να τονίσω τα εξή τρία. Συμφωνώ με την κυρία Γκόμες για τις ηλεκτρικές ε, διασυνδέσεις και τα δίκτυα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Υπάρχει ήδη συνεργασία αλλά θα πρέπει να ε, αυξηθεί. δεύτερο το εμπόριο δεν αφορά μόνο ε, αγαθά, υλικά αγαθά, εμπορεύματα, αλλά και υπηρεσίες. Ας μην έχουμε μονές με τα εμπορεύματα και θα πρέπει ε, σταδιακά, ε, με αμοιβαίο συμφέρον και με μελέτες αντικτύπου να ανοίξουν και αυτές οι αγορές. Αυτό δεν το λέγω μόνο, το έχω γράψει και σε μια τροπολογία στην υπαριθμόν 10 που ελπίζω να έχει την καλοσύνη να δεχτεί η συγκήτρια. Γιατί δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στις εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων. Και για να απαντήσω στον κύριο Κράισερ που μίλησε για τα τρόφιμα, βεβαίως δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο εξαγωγή τροφίμων. Γιατί το Μαρόκο και ε, την Ισία θα πρέπει να εξάγουν ε, ντομάτες και κολοκυθάκια. Γιατί δεν μπορούν να καλλιεργούν σιτάρι αντί να το εισάγουν από τη Γαλλία ή τις Ηνωμένε Πολιτείες. Γιατί έχουμε κολλήσει σε συγκεκριμένα εμπορεύματα που, ε, ε, και γεωργικά προϊόντα προς εξαγωγή και είναι εις βάρος της άλλης όχθης Μεσογείου. Θα πρέπει να είναι ευρεία η προσέγγιση της γεωργίας και όχι συγκεκριμένα τα προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται για εξάγονται στην Ευρώπη. Επίσης δεν με, με πειράζει ε, αν ε, χαρακτηρίζεται μόνο καλλιέργεια την ελιά στην Ανδαλουσία. Είναι πολύ ωραίο το τοπίο με τα ελαιόδεντρα, δεν με πειράζει. Για τις ε, κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις επίσης θα πρέπει να υπάρχει νομική ασφάλεια για να έρθουν οι ξένοι επενδυτές και να συνεισφέρουμε έτσι στην ευημερία. Δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα άνοιγμα εμπορικό για τα προϊόντα αλλά και για τις υπηρεσίες και μεταρρυθμίσεις, αυτό είναι το τρίτο, για να έχει εχέγγυα και ο ξένος επενδυτής να πάει να επενδύσει και να έχει μια ευημερία η περιοχή, πράγμα που όλοι επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την πολύ επικοδομητική αυτή συζήτηση και θα ήθελα ίσως να δώσω κάποιες απαντήσεις ήδη. Κατάρχά να πω εξ αρχής το εξής, ότι δεν μιλάμε για μια έκθεση, για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, δεν μιλάμε για νομοθετική έκθεση. Άρα, μπορούμε να μείνουμε σε πιο γενικό επίπεδο. Επίσης, ό,τι αφορά την ε, εμπορική συμφωνία με το Μαρόκο, την ψήφισε η Σχετική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και ξέρω ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες κάποιοι συνάδελφοι από μεσογειακές χώρες, αλλά αυτό είναι άλλη σελίδα. Νομίζω ότι εδώ σε μια τέτοια γνωμοδότηση δεν πρέπει να βάλουμε πάρα πολλά στοιχεία. Αυτό αφενός. Τώρα, κατά δεύτερον, στο κείμενο έχω αναφέρει τα κοινωνικά πρότυπα, την κοινωνική ευημερία, ότι όλα αυτά θα πρέπει να προωθηθούν, ότι επίσης οι περιβαλλοντικοί όροι θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τα κράτη της Μεσογείου να διαπράξουν τα ίδια σφάλματα που έχουμε διαπράξει κι εμείς. Ωστόσο, θεωρώ ότι θα πρέπει να υποδείξουμε και μπορούμε να υποδείξουμε ότι επικρατούν ε, δημοκρατικά πρότυπα και δημοκρατικές αξίες και κράτος δικαίου. Το ζήτησε η κυρία Κόμες ε, και το αναφέρω και εγώ στο κείμενο μου. Αν υπάρχει δημοκρατία και κράτος δικαίου, είναι αμοιβαία επωφελής οι σχέσεις μας και η διεξαγωγή εμπορίου. Αμοιβαία λοιπόν ανταλλαγή ε, υπηρεσιών, αγαθών, ενεργειακών πηγών. Ο Αυτά που θέλετε να αναφερθούν είναι βοήθεια για την αυτοβοήθεια ουσιαστικά. Είναι η μοναδική ουσιαστικά μορφή βοήθεια που λειτουργεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ύστερα κάποιοι συνάδελφοι ανέφεραν κάποιες μεταβατικές ρυθμίσεις, μα και αυτό αυτονόητο είναι. Αν κάναμε διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες συγκεκριμένα, ασφαλώς και θα ε, θέταμε μεταβατικές ρήτρε και προστασία για τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό αποτελεί ουσιαστικά μια σταθερά στην ευρωπαϊκή πολιτική. Μόνο που σε αυτό το κείμενο δεν ταιριάζει ουσιαστικά μια τέτοια αναφορά. Η αντίρρηση της κυρίας Κάκα, η οποία μίλησε για τον συνάδελφο Τα συμπεριλάβαμε αυτά. Είχαμε μια ανταλλαγή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα έχουμε ρυθμίσει αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που το επισημάνατε ωστόσο. Και ένα τελευταίο στοιχείο για τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, δεν ε, το ανέφερα συγκεκριμένα το θέμα αυτό, αλλά σε μία τροπολογία και, και αυτή της κυρίας Δεσσαρνές αναφέρεται με σαφήνεια ότι ότι θα πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες, οι γυναίκες και άνδρες. Νομίζω ότι αυτό επαρκεί. Αλλά αυτό φυσικά δεν μπορώ να το αποφασίσω εγώ μόνη μου, ίσως οι συνάδελφοι να έχουν διαφορετική άποψη. Νομίζω ότι επί της αρχής έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών έχει περάσει ήδη. Δεν είχαμε ευκαιρία να παρουσιάσουμε την έκθεση χωρίς τροπολογίες. Από όσο ξέρω θα ψηφιστεί την άλλη Δευτέρα η γνωμοδότηση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω τον Πρόεδρο με τη Σοφία που τον διακατέχει να μας υποβάλει μία πρόταση. Εγώ τι θα είχα υπόψη μου. Αν θέλετε να γίνει κάποια αλλαγή και θέλετε να μου την υποβάλλετε γραπτός, να την διαπραγματευτούμε, να την ε, επεξεργαστούμε ως προφορική τροπολογία. Ιδάλλως, ε, στα πλαίσια του κανονισμού δεν βλέπω κάποια άλλη δυνατότητα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά να παρακαλέσω τον Πρόεδρο να μου δώσει τη συμβουλή του. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Συγγήτρια. Στις 6 Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε και σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να εργάζεστε για τις συμβαστικές τροπολογίες αν μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι και προφορικά από τις 17 αυτές τροπολογίες. Αν μας ενημερώσετε γέρος και εμάς και τους και κάτι θα κάνουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Περνούμε στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης. Ευρωπαϊκή Ένωση, Αρμενία, Συμφωνία Σύνδεσης. Ο κύριος Τόμας Πιότρο Πορέμπα είναι, είναι συγητής μας. και η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου είναι αρμόδια, αλλά δήλωσε ότι δεν θα κάνει γνωμοδότηση, οπότε έχετε το ελεύθερο κύριε Πορέμπα απολύτω. Παρακαλώ, έχετε και το λόγο. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τι εργασίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Αρμενία. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έγγραφο του τελευταίου μήνε. Προετοίμασα όλες τις λεπτομέρειες. Επισκέφθηκα τον Αγκόνο Καραμπάχ στην Αρμενία συνομίλησα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, με τον πρόεδρο ε, της χώρας, με τον πρωθυπουργό, με εκπροσώπους των μη κυβερνητικών οργανώσεων, προκειμένου να προετοιμάσω το, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έκθεση αυτή για την κατάσταση στην Αρμενία και στην όλη περιφέρεια. Προκειμένου η έκθεση λοιπόν αυτή να είναι ολοκληρωμένη και αντικειμενική. Μια έκθεση η οποία θα αποτυπώνει πραγματικά την κατάσταση όσο έχει στην Αρμενία την πολιτική κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση και θα ήθελα να εξετάσουμε και την περιφερειακή κατάσταση στο σύνολό τη, προκειμένου να εγκριθεί αυτή η έκθεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμβάλλει στη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊ... μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αρμενίας. Επίσης, ε, έλαβα υπόψη διάφορα ζητήματα, τα οποία Φαίνεται ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση στην Αρμενία, αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να χρήζουν περαιτέρω βελτίωση. Όλα αυτά λοιπόν τα έχω αναφέρει. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι προσπάθησα να συμπεριλάβω τις απόψεις όλων και να πω ότι ειλικρινά θα χαρώ να ακούσω τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας προκειμένου να ενισχυθεί η έκθεση, να βελτιωθεί Και αντιλαμβάνομαι ασφαλώς ότι διάφορα ζητήματα μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Σε αυτά συγκαταλέγεται και η καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία θα πρέπει να γίνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Προκειμένου οι παλιές ε, πρακτικές της πολιτικής θα πρέπει να αλλάξουν σε ό,τι αφορά τα θέματα, τα δικαστικά και τις ανεξαρτησίες των δικαστικών αρχών. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει βελτίωση, θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση θεωρώ σε ό,τι αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα την ελευθερία έκφρασης του Κοινοβουλίου και σε ό,τι αφορά τις μόνιμες επιτροπές πιο ειδικά. Να σας υπενθυμίσω ωστόσο ότι κάποια στοιχεία έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση της Αρμενίας, έχουν αποδεχτεί όλες αυτές τις ε, απαιτήσει έχουν προσπαθήσει να προσαρμόσουν τις αξίες στις δικές μας αξίες και αυτό κατέστησε σαφές ε, στις επαφές μου με τις ε, κρατικές αρχές όλες με διαβεβαίωσαν ότι ο στόχος της ε, κατεύθυνσης της Αρμενίας είναι η Ευρώπη. Θέλουν να μεταρρυθμιστεί το κράτος τους, θέλουν να βρουν λύσεις οι οποίες θα προσεγγίσουν την Αρμενία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιθυμούν να διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο η Αρμενία στην περιφέρεια, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιφέρεια. Άρα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στην Αρμενία το γεγονός ότι έχει ήδη ολοκληρώσει και κλείσει πολλά κεφάλαια, για παράδειγμα την αστυνομική μεταρρύθμιση. Στο κράτος αυτός, αυτό ο αριθμός των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να επισημανθεί, να επισημανθεί όπως ε, επίσης η ανάπτυξη του γραφείου του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά καταδεικνύουν πόσο σοβαρά παίρνει η Αρμενία τα ζητήματα αυτά. Σε ό,τι αφορά επίσης τις συμφωνίες ευκόλυνσης της χορήγησης θεώρησης, και σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή, σε ό,τι αφορά θέματα ελεύθερης ζώνης εμπορίου. Όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και πολλά μπορούμε να πετύχουμε στο Κοινοβούλιο, αλλά ήδη έχουν επιτευχθεί και πολλά από αυτά τα στοιχεία. Θα ήθελα η έκθεση αυτή να αποτελέσει και ένα έγγραφο το οποίο θα βοηθήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Αρμενία στην περαιτέρω μεταρρύθμιση και ενίσχυση του κράτους της Αρμενίας. Ασφαλώς ε, και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλά ευαίσθητα και ακαθόδη ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα α, σκεπάσουμε, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Τον Αγκόρνο Καραμπάχ, για παράδειγμα. Μετέβησα στον Αγκόρνο Καραμπάχ, λοιπόν, και καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει εκεί, πώς έχει το συνολικό πλαίσιο και η κατάσταση εκεί. Θα ήθελα ωστόσο να σας παρακαλέσω, συνάδελφοι, η έκθεση αυτή σε ό,τι αφορά την Συμφωνία Σύνδεσης. Να μην περιοριστεί. Να μην συνδεθεί καν με το θέμα του Νεγκόρνου Καραμπάχ. Άρα, να ακούσω τις προτάσεις σας, ευχαριστώ και ως εισηγητής πρέπει να σας πω, θα εμείνω στο ότι το θέμα του Ναγκόνο Καραμπάχ θα πρέπει να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της ομάδας Μίνσκ. Προκειμένου να προκύψει τελικά ένα έγγραφο το οποίο δεν θα ανοίξει τα κουτί της Πανδώρας εκ νέου. Αυτό θα ήθελα να το αποφύγω. Δεν θα ήθελα να επηρεάσουν αυτά την έκθεσή μου. Ασφαλώς και πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και πάντα σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ο εισηγητής ουσιαστικά ακούει αυτά που έχουν να πούν οι εκπρόσωποι των διαφόρων ομάδων. Άρα δεν θα μακρηγορήσω. Να ακούσω τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και να ακούσω ιδιαίτερως και τα σχόλια των σκιωδών εισηγητών. και θα ήθελα η έκθεση αυτή για την Αρμενία να είναι αντικειμενική και να λάβει υπόψη και τις ε, ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αρμενίας που είναι ειλικρινής χωρίς να ξεχνάμε και να κρύβουμε ότι χρειάζονται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας. Ο κ. Κόβαλτσεφ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Στα αγγλικά θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Πορέμπα ε, για την ε, παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης που είναι πάρα πολύ αντικειμενική και ισόρροπη. Πριν μπω στα θέματα της Συμφωνίας Σύνδεσης, θα ήθελα, μου επιτρέπετε, να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Όταν συζητούμε για θέματα Αρμενίας Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην δίνουμε επιχειρήματα επιρομαχικά στη συζήτηση ε, στη μία την άλλη πλευρά. Πράγμα που είχε συμβεί δυστυχώς στο παρελθόν με μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα σημεία G και H μπαίνω πρώτα στην παγωμένη σύραξη το καθόθε ζήτημα. Συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά στο σημείο G ε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέτε για την Αρμενία. Δεν ξέρω αν είναι θέμα μετάφρασης. Στο G, στο Z και για την ομάδα του Μίνσκ. Θα πρέπει να βρεθεί ε, μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Στο μικρό ζήτα, λοιπόν, στα ελληνικά, εκεί λέει για όλη την επικράτεια της Αρμενίας. Αυτό είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Επίσης, ε, μπορεί μια τέτοια συμφωνία να εφαρμοστεί με κλειστά τα σύνορα και πρόβλημα στη διαμετακόμιση. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την Τουρκία και την Αρμενία, περισσότερο την Τουρκία και λιγότερο την Αρμενία, να ανοίξουν τα σύνορα. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη πολιτική γειτονία, λεγόμενη προσέγγιση more for more, περισσότερα με αντάλλαγμα και περισσότερα. Ε, οι μεταρρυθμίσεις που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν την Αρμενία και θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ε, ε, διαδεδομένη σύλλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς την Αρμενία και τον αρμενικό λαό. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ε, ότι χαίρομαι για την έναρξη των διαπραγματεύσεων και τη διαδικασία απελευθέρωση θεώρηση διαβατηρίων. Θα ήθελα να εθαρρύνω επίσης την Αρμενία να επιταχύνει την αναγνώριση του καθεστώτος στον Ρωμά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και να καταπολεμήσει περισσότερο τη διαφορά, όπως είπε και ο Τέλος, κάτι που είναι πολύ σημαντικό φέτος, είναι οι εκλογές του Μαΐου που θα πρέπει να γίνουν ε, απρόσκοπτα και με ε, ελεύθερο τρόπο και θα είναι μια δοκιμασία για τη ε, δημοκρατία στην Αρμενία. Ελπίζω να ακολουθήσουν το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης εισηγητής από τους σοσιαλδημοκράτες. Σπάνια ε, ο σκιώδη προσθέτω κάτι σε μια έκθεση. Είναι πάρα πολύ επαγγελματική και πολύ αντικειμενική η έκθεση προκειμένου να μην προκύψει καμία σύγκρουση. Γίνεται παράλληλη προετοιμασία των διεκθέσεων για, το, για την Αρμενία και για το Αζερβαϊτζάν. Αυτό είναι σωστό. Γι' αυτό λοιπόν έχω να προσθέσω τα εξή. Ε, Έναξη παράθεσης οι διαπραγματεύσεις για το πρόβλημα των Αγκόρνων Καραμπάχ θα πρέπει να διεξαχθούν πιο εντατικά. Γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των πολιτών του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Η δίκαιη και αμοιβαία ε, ισότιμη λύση θα δώσει κίνητρο στην οικονομική ε, ανάκαψη των χωρών. Τέλος παράθεσης. Γι' αυτό θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να προωθήσουμε την ε, εμπορική συμφωνία. Και τέλος θα ήθελα συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Παρέμα για την εξαιρετική έκθεση. Όταν δεν έχει τίποτα να προσθέσει ένας σκιώτης εισηγητής, πραγματικά πρόκειται για πολύ επιτυχημένη έκθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και από πλευρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Πορέμπα για την πάρα πολύ συνοπτική έκθεση που συμπεριλαμβάνει τα πιο σημαντικά στοιχεία. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα εξ αρχής. Καταρχάς, να κάνω μια ερώτηση προς τη γραμματεία. Γιατί ε, έχουμε τόσο σύντομη χρονική προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Μεθαύριο, δύο μέρε μόνο. Και η έκθεση θα ψηφιστεί στην Επιτροπή στα τέλη Φεβρουαρίου από τις 19 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, όπως ξέρετε, μια αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ θα μεταβεί στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν, μεταξύ άλλων. Άρα νομίζω ότι σκόπιμο θα ήταν να έχουμε μεγαλύτερη προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. Ξέρω ότι ίσως να αντιμετωπίσει δυσκολίες ε, η γραμματεία, αλλά να έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί η τελική ψηφοφορία τελικά στην Ολομέλεια θα είναι στη δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου. Ε, άρα νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα να μεταβούμε στην περιοχή και τα συμπεράσματά μας να τα συμπεριλάβουμε και στην ε, έκθεση. Αυτό το απευθύνω ως έκκληση και στην γραμματεία αλλά και στον εισηγητή. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι όντω είναι καλό το γεγονό ότι γίνεται ταυτόχρονη επεξεργασία και των δύο εκθέσεων. Όπω είπε και ο κ. Κόβατσεκ, θα πρέπει να καταστήσουμε σαφέ ότι θα είναι ίση η αντιμετώπιση προκειμένου να μην προκύψουν προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν, αν θέλετε, επιχειρήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ο ένας κατά του άλλου για τις τροπολογίες τώρα. Θα τις κάνουν τις τροπολογίες τις ίδιες και για την έκθεση για το Αζερμπάιτσαν. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που ήθελα να αναφέρω. Ότι όντως υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα και έγκυται στο ότι και οι δύο χώρες αποτελούν τμήμα της ανατολικής γειτονικής σχέσης, αλλά ουσιαστικά ε, βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση μία με την άλλη. Αυτό νομίζω αποτελεί πρόβλημα και για μας σε ό,τι αφορά την διαπραγμάτευση και τις συζητήσεις ε, και με τις δύο χώρες. Το είδαμε και στη Γυρονέστ. Θα πρέπει λοιπόν να καλέσουμε τις δύο χώρες να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ότι η Συμφωνία Σύνδεσης σημαίνει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Σε ό,τι αφορά την Αρμενία θα πρέπει να ζητήσουμε ε, η παναχώρηση των αρμενικών στρατευμάτων, γιατί αν προκύψει σχετική συμφωνία με τις δύο αυτές χώρες, θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις πρόοδος στον τομέα της ειρηνευτικής πολιτικής. Ένα άλλο σημείο σε ό,τι αφορά τις εκλογές, τις επερχόμενες εκλογές το Μάιο του 2012 στην Αρμενία. Θα πρέπει νομίζω να καλέσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να διασφαλίσουν την πρόσβαση στα μέσα για την προετοιμασία της προεκλογικής εκστρατείας σε ό,τι αφορά τους προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τώρα και γενικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε τέτοιες αναφορές. Επίσης, να αναφερθεί και το θέμα του περιβάλλοντος. Υπάρχει ένα περιφερειακό γραφείο, κέντρο για το περιβάλλον, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι αναφορές. Όχι σε ό,τι αφορά μόνο την Αρμενία και το Ζαρμπαϊτζάν, αλλά και τη Γεωργία και όλη την περιφέρεια. Πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν. Δεν σημαίνει το γεγονό ότι επειδή υπάρχει ένα πλησίραξη σε μια περιφέρεια ότι θα πρέπει να παραμεληθούν τα θέματα του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να τα επισημάνουμε όλα αυτά και μάλιστα εγκαίρως. Α, και ο κ. Κοβατσέκ επίσης αναφέρθηκε στο ζήτα, το μικρό ζήτα, για την αναφορά σε όλη την επικράτεια της Αρμενίας. Εδώ θα καταθέσω μια τροπολογία για να σβηστεί, να διαγραφεί αυτή η πρόταση. Να αναφερθεί μόνο ε, η συμφωνία του ΟΗΕ του Ελσίνκη να μην προκληθεί όμω ε, σύγχυση και παρανόηση με την αναφορά αυτή σε όλη την επικράτεια της Αρμενίας. Κάτι άλλο και για τις δύο εκθέσει. Θα πρέπει να το επικρίνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι και στις δύο χώρες ε, είναι έντονη η... ο εξοπλισμός γενικότερα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε, θα πρέπει να αναφερθεί. Κάτι άλλο ως ε, πράσινη πολιτικός. Θα καταλάβετε ασφαλώς πόσο σημαντικό είναι για μας να παραπληστεί το πυρηνικό εργοστάσιο του Μετζαμόρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι και προσβλέπω στις αντιπραγματεύσεις μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαρλάκη. Thank you. Uh, this is an initial discussion. Σας ευχαριστώ. Είναι μια πρώτη συζήτηση για αυτές τις δύο συμφωνίε και εκτιμώ ιδιαίτερω το ότι τα συζητάμε από κοινού. Επίσης εκτιμώ την πρόταση όπως διατυπώθηκε από την εισηγήτρια, είναι καλή, ισορροπημένη και διέπεται από καλές προθέσεις. Επίσης συμφωνώ με άλλους συναδέλφους ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ε, σύγκρουση Ναγκόρνο Καραμπάχα όταν συζητάμε μια τέτοια συμφωνία σύνδεση με αυτές τις δύο χώρες. Και κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στη διαπραγμάτευση μιας ε, λύσης. Ακόμα και αν ε, καταρχήν δεν είμαι υπέρ της ε, θέσεις όρων σε οτιδήποτε, σε αυτή την περίπτωση πιστεύω πως μία σύνδεση ανάμεσα στη Συμφωνία Σύνδεσης και της προόδου προς μια ειρηνική λύση στο θέμα του Ναγκόρνου Καραμπάχ νομίζω θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τα όσα ήδη κάναμε ως ε, κοινοβούλιο για την έκθεση για την στρατηγική για τον Νότιο Κάφκασο πέρσι τον Απρίλιο, καθώς και επίσης ε, με σε βασικές αρχές ε, ψήν ψηφίσματα του ΟΙΕ. Η πρότασή μου δεν είναι τροπολογία ακόμη, δεν, είναι μια, προ, πρόταση προ-τροπολογίας και ζητώ από τον συνάδελφο να τη λάβει υπόψη, δηλαδή να συνδέσουμε τις δύο συμφωνίες με, τρεις, με τρία σημεία. Την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης και πρόληψης ε, περιστατικών για τις δύο χώρες, την απόσυρση των αρμενικών ε, δυνάμων από τα κατεχόμενα εδάφη του Αζερβιτζάν και των Αγκόρνο Καραμπάχα και την ε, δημιουργία μιας ε, γνήσιας ε, δύναμης διατήρηση της ειρήνης στο ε, περιοχή αυτή. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να το συζητήσουμε. Είμαστε στις αρχές της συζήτησης στην σοσιαλιστική ομάδα και θα ήμουν ευτυχής αν συνάδελφοι από άλλες ομάδες εξέφραζαν την θέση τους, τη γνώμη τους για αυτήν την προ τροπολογία. Σα ευχαριστώ πολύ, Έχω μία ερώτηση και δύο σχόλια. Η αστυνομία της Δημοκρατίας της Αρμενίας επιτρέπεται τώρα να ελέγχει ε, όλα ε, τα σώματα που διενεργούν έρευνες αλλά εκφεύγει του ελέγχου η ίδια αστυνομία μετά τη δολοφονία του Υπουργού Εσωτερικών. Και ρωτώ τον εισηγητή, πού, ποιος είναι ο έλεγχος και η εποπτεία υπάρχει τέτοιος, ε, υπάρχει κάποιο υπουργείο ή το κοινοβούλιο που να ελέγχει την αστυνομία στην Αρμενία. Και τι γίνεται με όλα τα διοκτικά σώματα. Γενικότερο σχόλιο. to οι προσπάθειες αποφυγής σαφούς θέσεως ή οποιασδήποτε λήψης θέσεως για ένα παγωμένο, παγωμένη σύραξη και ε, δεν κατανομάζουμε την αιτία ε, του κακού, τη βασική αιτία στο Νότιο Κάφκασο που είναι ότι κατέχεται μια επικράτεια από μια γειτονική χώρα. Γι' αυτό έχω κάνει κάποιες μικρές τροπολογίες τουλάχιστον να ε, σημειώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και τι θα μπορούμε να πούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην ντροπιαστούμε. Θα μας σώσει η έγκρισή τους και παρακαλώ να μην τις απορρίψετε. Και τελευταίο σχόλιο. Το να συνδεθούν οι δύο συμφωνίες σύνδεσης, ακόμα και οι τρεις για τις τρεις χώρες του Νοτιού Καυκάσου, είναι αντίστοιχο ε, με μια πάρα πολύ έντεχνη παγίδα. Δηλαδή πώς να μπλοκάρουμε και τα τρία αυτά σε ένα για να μην μπορέσει να προχωρήσει καμία από τις συμφωνίες σύνδεσης. Παρακαλώ να το αποφύγουμε. Σας ευχαριστώ. Thank you, Chairman. First Uh, just as it was Κύριε Σκυρίλοφ, ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι όπως είπαν και οι συνάδελφοι είναι καλό το γεγονός ότι συζητάμε παράλληλα τις δύο αυτές εκθέσεις. Και είναι επίσης ε, σωστό ότι προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ισορροπή και μια ίση αντιμετώπιση, φυσικά επικεντρωνόμενη στο στόχο μας. Ο στόχος λοιπόν είναι η πιο ενεργή συμμετοχή, η πιο ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα θέματα αυτά τα μεγάλα στρατηγικά συμφέροντα της ε, Ένωσης στην περιφέρεια αυτή είναι να υπάρχει σταθερότητα και ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν ε, προσέξατε την ε, πέρσινη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αναφέρεται ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις που επηρεάζουν ε, διάφορες γειτονικέ χώρες και αναφέρεται ρητά ο Νότιο Κάφκασο, αποτελούν μια σημαντική απειλή για την ασφάλεια όλη της περιφερεια και για τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζονται από την αστάθεια αυτή που επικρατεί. Άρα θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή Μεν για όλη την έκθεση η οποία είναι ισόρροπη αλλά παράλληλα θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν μπορούμε απλά να μην κάνουμε τίποτα α, για αυτή τη συνεχιζόμενη σύγκρουση που σε λίγο θα κλείσει 20 ετία. Θα πρέπει να λάβουμε τις ευθύνες μας. Νομίζω ότι η επερχόμενη αυτή αποστολή της Επιτροπής ε, ε, Εξωτερικών Υποθέσεων στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Γιατί και το κοινοβουλίο μας δεν μπορεί να μένει αμέτωχο. Είναι στο συμφέρον μας να αντιδραματίσουμε ρόλο σημαντικό να δημιουργήσουμε τους όρους για την ανάπτυξη ε, εμπιστοσύνης, να μιλήσουμε με τα κοινοβούλια και των δύο χωρών, να είναι επικοδομητικές οι συζητήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Αρλάκη. Θα πρέπει η διαδικασία αυτή να συνδεθεί με την όλη αξιολόγηση της ε, Αρμενίας και του Ζερβαϊτζάν σε ό,τι αφορά τη μελλοντική συμμετοχή και συμφωνία σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τηρήσουμε πολύ λεπτές ισορροπίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες ιδέες που αναφέρονται στην έκθεση, πολύ σωστές. Νομίζω ότι θα πρέπει και στις δύο χώρες να επικεντρωθούμε, ιδιαίτερα επειδή έχουμε τις επερχόμενες εκλογές, να επικεντρωθούμε λοιπόν στην διεξαγωγή σωστών εκλογών στην περιφέρεια. Και μια και η Επιτροπή ΑΦΕΤ θα, θα πάει για τι εκλογέ στην Αρμενία, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και στην τελευταία μου επίσκεψη στην Αρμενία ήταν μεγάλε οι δεσμεύσει. Ε, από πλευρά τη κυβέρνηση και του Προέδρου για την διεξαγωγή δίκαιων εκλογών αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το ενισχύσουμε στην έκθεση σε ό,τι αφορά την τεχνική αρρωγή που θα χορηγήσουμε στις χώρες αυτές, ιδιαίτερα στην Αρμενία τώρα στις επερχόμενες βουλευτικέ εκλογές. Αυτά θα πρέπει ασφαλώς ε, η αρρωγή αυτή να προκύψει και από τους άλλους δημοκρατικούς εταίρους, όπως το ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το καθεξής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Chair. I don't want to repeat what... Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Φαίνεται να είναι ευρία η συνένεση, λέει ο κύριο Βίγκενιν, μεταξύ των συγητών και των σκιωδών. Συγχαρητήρια για την έκθεση. Επιτρέψτε μου να πω το εξή. Θα πρέπει να είμαστε βεβαίω πάρα πολύ προσεκτικοί ε, σε αυτή την ιδέα, να συνδέσουμε δηλαδή το θέμα του ορεινού Καραμπάχ ε, με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης Συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά να μην το παρακάνουμε, δηλαδή να μην συνδέσουμε την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την επίλυση αυτής της σύγκρουσης. Θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Ξέρουμε από την εμπειρία μας ότι αυτό το θέμα είναι από μόνο του σε θέση να οδηγήσει σε εμπλοκή την όλη διαδικασία. Προσοχή λοιπόν. Επίσης είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο χώρες και το γενικό περιβάλλον στο Νότιο Κάφκασο να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες σύνδεσης, να τις επιταχύνουμε και ταυτόχρονα μάλιστα να προχωρούμε και κάπως να συνδέσουμε και τις δύο χώρες στην ευρωπαϊκή προοπτική για να τη χαρακτηρίσω έτσι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι προς το παρόν τουλάχιστον αυτό το θέμα φαίνεται να είναι πιο εκκληστικό και πιο σημαντικό για την Αρμενία η οποία προοδεύει ταχαίως τις διαπραγματεύσεις. Από την άλλη, από ό,τι φαίνεται το Αζερμπαϊτζάν, πώς να το πω, δεν έχει ξετρελαθεί από το ενθουσιασμό του και αν μιλούμε για άσκηση πίεσης και προς τις δύο πλευρές θα πρέπει να τα λάβουμε και αυτά υπόψη. Και τέλος ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Η πρώτη επίσημη αντιπροσωπεία φέτος ε, της Επιτροπής μας θα μεταβεί στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να αφήσουμε λίγο περισσότερο χρόνο για τις τροπολογίες και αυτό θα μας βοηθήσει να μελετήσουμε προσεκτικά τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε στις τροπολογίες μας για να συνδεθεί ε, αυτό το θέμα με τον ε, Ναγκόρνο Καραμπάχ και ελπίζω να υποβληθεί με υπογραφές βουλευτών από τις σημαντικότερες πολιτικές ομάδες για να έχει και μεγαλύτερη ισχύ. Ενημερωτικά, τέλη Φεβρουαρίου, μία από τις επιτροπές της Euronest θα συνεδριάσει στην Αρμενία αμέσω μετά τη δική μας επίσκεψη. Ελπίζω αφενός να συμβάλλουν αυτά στα όσα σας είπα, αλλά και η δική μας ε, αντιπροσωπεία στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν και ε, η συνεδρίαση της Επιτροπής στο Γερεβάν θα μας βοηθήσει να ανταλλάξουμε και απόψεις και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους ότι είναι καλό να συζητήσουμε ταυτόχρονα τις δύο εκθέσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ε, παρουσιάστηκε μια άλλη έκθεση για το Αζερβαϊτζάν και μετά να έχουμε μια κοινή συζήτηση. Ε, πάση περιπτώσει. Στην ουσία συζητάμε τις δύο εκθέσεις τώρα, οπότε θα κάνω και εγώ την εξή παρατήρηση. Το βασικό μήνυμα είναι το, η ευρωπαϊκή προοπτική και για τις δύο χώρες. Είναι προς το συμφέρον μας. Είναι ο μόνος τρόπος για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αναφέροντας το πρόβλημα του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Είναι ένα τόσο γνωστό θέμα και τόσο πολύ συζητημένο που δεν θα πρέπει να φοβηθούμε να το αναφέρουμε. Με πολύ ξεκάθαρο τρόπο σε αυτές τις εκθέσεις. Μα αυτό είναι ο ρόλο μα, αγαπητοί κύριοι. Αυτό είναι ο ρόλο του Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνω πω οι διπλωμάτε μπορεί να μην τα λένε τόσο έξω από τα δόντια, αλλά εμεί πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί διαφορετικά δεν βοηθάμε στη λύση του προβλήματο δεν θα πρέπει να Προσε... Δεν θα πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή του, του, της διατύπωσης, αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματά μας. Νομίζω πως δεν αρκεί να ε, δηλώνουμε υποστήριξη στην ε, ομάδα Μίνσκ, του Μίνσκ, αλλά μέχρι στιγμής δεν είχε αρκετά μέσα στη διάθεσή της για να αποδώσει σε ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα. Είναι πολιτικής φύσης πρόβλημα, θα πρέπει ε, έτσι να το αντιμετωπίσουμε και νομίζω αν πούμε απλά εντάξει είναι δουλειά της ομάδας του ΜΙΣΚ κατά κάποιο τρόπο δεν είμαστε αξιόπιστοι. Νομίζω πως υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν πρέπει να τα αποφύγουμε. Ας πούμε το δικαίωμα των προσφύγων να επανέλθουν και στα σπίτια τους. Είναι ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Ισχύει για τους πρόσφυγες που έφυγαν από το Ναγκόρνο ο Καραμπάχ επειδή ήταν Αζέρι και για τους Αρμένους που έφυγαν από την Πακού επειδή ήταν, είναι Αρμένοι. Είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να το τονίσουμε εμείς οι ε, βουλευτές. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε τη λύση του προβλήματος του Ναγκόρνου Καραμπάχ μέσα στο πνεύμα του διεθνούς δικαίου. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο στις διεθνείς ε, σχέσεις παρά η διεθνή νομοθεσία, το διεθνέ δίκαιο. Και αυτό φυσικά ισχύει και για την ε, απόσυρση των στατευμάτων από τα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη. Ε, αυτό που κατά τη γνώμη μου λείπει από αυτή την έκθεση είναι ότι θα πρέπει να ε, μιλήσουμε για τους, στους αρμένιους φίλους μας, αν θέλουμε το καλό τους, ε, να μιλήσουμε και για τη ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Αρμενία που βλάπτει την υπόθεση, το καθιστά ακόμα πιο περίπλοκο και ζημιώνει και τη θέση της Αρμενίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος συζητητής, ο κύριος Πορέμπα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο ε, κατά τη συζήτηση της εκθέσεώς μου. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφερθώ σε μερικά από τα όσα είπατε. Συμφωνώ, κυρία Λούνατσεκ, και με τον κύριο Κόβαλτσεφ. Για το σημείο Ζ έχω και σχετική τροπολογία. Είμαι απολύτως της απόψεως να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και συμφωνώ ε, και για τα τουρκο-αρμενικά σύνορα έχω σκεφτεί να προετοιμάσω και εγώ μια τροπολογία για να διασκεδάσουμε όλες τις αμφιβολίες και τους φόβους ε, του βουλευτού. Λοιπόν, να απαντήσω τώρα στον κύριο Λαντσπέργης. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα πρέπει να το ελέγξουμε ε, και να το επαληθεύσουμε. Αναφέρθηκα σε κάποιες μεταρρυθμίσεις και θεσμικές και γενικότερες. Σας υπόσχομαι ότι θα ε, το κάνω οπωσδήποτε, θα επαληθεύσω την κατάσταση εκεί ως ε, εισηγητής. Για το Ρινό Καραμπάχ κατανοώ τα επιχειρήματα που λέγουν ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε περισσότερο σε αυτή την υπόθεση και να μιλάμε ξεκάθαρα. Πιστέψτε με όμως, γιατί εγώ έχω ζήσει λίγο στην περιοχή εκεί. Έκανα επισκέψεις και στην Αρμενία. Και η είναι πολύ μεγάλη. Τα συναισθήματα βράζουν. Είναι πολύ φορτισμένη η κατάσταση και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, και στη διατύπωσή μας για τη Συμφωνία Σύνδεσης, γιατί δεν έχω την εντύπωση ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε σε θέση να λύσουμε ε, αυτή την υπόθεση, αυτό το ζήτημα και τη σύραξη. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιγράψουμε την κατάσταση ειλικρινά, ενδεχομένω να ε, υποβάλουμε και συστάσει για τα μελλοντικά, τα επόμενα βήματα, αλλά για μας θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λύσουμε ε, τη διαφορά αυτή. Παρακαλώ να με καταλάβετε. Η έκθεση αφορά την Αρμενία. Βεβαίως δεν μπορεί να αφήσει κανείς τελείως έξω τον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά Συμφωνώ με τους ηγητές, θα πρέπει να επιλέξουμε πάρα πολύ προσεκτικά τη διατύπωσή μας για να έχουμε πραγματικά ουσιαστικά αποτελέσματα και να περιγράψουμε την κατάσταση όπως έχει. Εγώ είμαι πρόθυμος να το κάνω, αν θέλετε, αλλά θα παρακαλούσα έντονα να μην τον περιορίσουμε ε, το θέμα μόνο ε, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στην έκθεση αυτή. Βασικός στόχος είναι να αντικατοπτριστεί αντικειμενικά η κατάσταση στη χώρα. Τι θέλει η Αρμενία, τι προσδοκίες έχει, πώς θέλει να λειτουργήσει στο εσωτερικό της Ευρώπης και ε, τι γίνεται με τα κριτήρια και ε, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Εγώ θα επιθυμούσα η έκθεση αυτή να συνεισφέρει προς αυτή την κατάσταση. Να πούμε ε, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πώς φροντίζει να βοηθήσει την Αρμενία. Ελπίζω να είμαστε σε θέση να το διατυπώσουμε έτσι με ένα επικοδομητικό τρόπο Προσβλέπω στη συνεδρίαση με τους κοιόδης ηγητές και δεν μπορώ παρά να επαναλάβω ότι είμαι πρόθυμος να δεχθώ όλες τις συστάσεις και τις προτάσεις σας για να βελτιωθεί, να υποστηριχθεί η έκθεση. Έτσι ώστε να μπορέσουμε και να ψηφίσουμε γνωρίζοντας ότι έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να είναι η έκθεση καλή και να εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές δηλαδή και την Αρμενία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Λατσπέργης, ένα μικρό σχόλιο. Ακούω για την πρόοδο που λέτε, για τις προσδοκίες, για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ωραία όλα αυτά. Αλλά πρόσφατα είπε ο Δημήτρη Μετβέντεφ σε κάποιους δημοσιογράφους στο Καζάν ότι έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Αρμενία, η Ρωσία. 80% της βιομηχανίας της Αρμενίας ανήκει σε ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις. Μεγάλη πρόοδος, ναι, 20% είναι το υπόλοιπο ε, της πρόοδου. Μας ικανοποιεί με τον ίδιο τρόπο και το χαιρετίζουμε. Σε ευχαριστώ. Από αυτό μπορούμε να εξεγάγουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, αλλά θα δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Από ό,τι άκουσα, διάφοροι συνάδελφοι ζήτησαν να παραταθεί η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Ε, σκόπιμο είναι, θεωρώ, προκειμένου αυτές οι διεκθέσεις για την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να ψηφιστούν τον Απρίλιο και ε, να μετατεθεί η κατάθεση, η ημερομηνία για τις τροπολογίες 28 στην 28 Φεβρουαρίου, μετά την ε, αντιπροσωπεία, δηλαδή μετά την επιστροφή της αντιπροσωπείας. Αφού θα πάει που θα πάει η αντιπροσωπεία. Είναι καλή αυτή η πρόταση. Συμφωνείτε να αλλάξει έτσι το χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στο σημείο 9, στην έκθεση της κυρίας Γιάντεμακη. Σας ευχαριστώ πολύ. που είσαστε εδώ για να μας παρουσιάσετε για την έκθεση και τη Συμφωνία Σύνδεσης με το Αζερβαϊτζάν. Μιες, σας ευχαριστώ. Το Αζερβαϊτζάν πρόσφατα κάλυψε το στήλος των εφημερίδων. Ήταν μάλιστα αποτέλεσε και ένα από τα θέματα στο Νταβός. Η οικονομία του αναπτύσσεται και αυτό ενδιαφέρει πολύ τη Δύση. Η πετρελοβιομηχανία επίσης έχει αναπτυχθεί πολύ, καθώς και η υπόλοιπη οικονομία. Προχωρούν, αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από ότι εμείς. Μάλιστα, η βαθμολογία του ως προς την πιστοληπτική του ικανότητα έχει αυξηθεί. Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει από τη δικιά μας γειτονιά. Οπότε είναι πολύ θετικό να, να, ξεκινάμε διαπραγματεύσεις σύνδεσης με μια τέτοια χώρα. Έχουμε επισκεφθεί αυτή τη χώρα και είχαμε επαφές με τον Επίτροπο Κάλας και θέλουμε Μάλλον και από ό,τι μαθαίνουμε, το Αζερβαϊτζάν θέλει να διευρύνει τις αγορές με τις οποίες ε, συνεργάζεται και μάλιστα θέλουμε μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης να διαπραγματευτούμε και μια ειδική συμφωνία για την ενέργεια ως μέρος ε, της ευρύτερης συμφωνίας. Δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει βέβαια τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές καθ' αυτές. Δεν είναι λοιπόν απλά οικονομικό το ζήτημα, όπως αναφέρθηκε στον Ταβό για προφανείς λόγους, αλλά είναι και ένα θέμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, όπω όλοι γνωρίζουμε. Σε αυτούς τους τομείς έχουν πολλά ακόμα να γίνουν στο Αζερβαϊτζάν. Κάποια πράγματα έχουν γίνει όσον αφορά την ελευθεροτυπία, την ελευθερία λόγου, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και η αντιπολίτευση, η ΜΚΟ, πρέπει να είναι πιο ελεύθεροι, να είναι σε θέση να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι ε, απόδειξη δημοκρατίας και φυσικά είναι και μέρος των δικαιωμάτων του λαού του Αζερβαϊτζάν, ελευθερία λόγου, ελευθερία άποψης και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτές τις πτυχές όταν αναζητούμε λύσεις ε, και διαπραγματευόμαστε σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν. Πρόεδρε, εγώ έχω να σχολιάσω τα όσα υπόθηκαν σε σχέση με την Αρμενία. Στην προηγούμενη έκθεση, λόγω της ε, σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι πρόβλημα. πρέπει κανείς να βλέπει επιφυλακτικά την ομάδα του μίνς και δεν έχει επιτευχθεί τίποτα, δεν έχει υπάρξει πρόοδος. Όμως, Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν υπήρξε εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ομάδα Μίνσκ και Γαλλία, η Ρωσία και η ΕΠΑ ήταν παρούσες. Δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσία εκπροσώπηση της Ένωσης και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά παράξενο για να το πω έτσι ήπια. Ωστόσο, έχουμε συχνά μιλήσει για την ανάγκη εξέβρεσης λύσης για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. και συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή, τον κύριο Πορέμπα, ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι Μπορεί να σκεφτόμαστε στο Κοινοβούλιο ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξέβρεση λύση σε αυτή την ε, σύγκρουση. Η Ένωση δεν αποτέλεσε ποτέ μέρος της λύσης σε αυτά τα προβλήματα. Και αυτό είναι μια δυσκολία που πιστεύω πρέπει να την εξετάσουμε. Συμφωνώ με τα όσα είπατε για το άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας. Είναι δύσκολο να το λύσουμε αυτό μέσω μιας ψηφοφορίας θα πρέπει να είμαστε, ε, θα είμαστε διχασμένοι. Και κανένα μέρος δεν φαίνεται να θέλει να προσεγγίσει το άλλο. Πρέπει αυτό να το δεχτούμε και να δεχτούμε ότι η Ένωση στην ουσία έχει μείνει στην άκρη. Ο κύριος Λούνατσεκ ανέφερε, η κυρία με συγχωρείτε, Λούνατσεκ ανέφερε ότι θα πρέπει να επικρίνουμε αυτού του αγώνα εξοπλισμών μεταξύ των δύο χωρών. Είναι αλήθεια ότι πολλοί πόροι ε, τους έχουν ε, πάει στην αγορά όπλων, πράγμα το οποίο δεν έχει βοηθήσει την ευημερία των λαών. Ο κ. Κόβατσεφ και άλλοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Και εγώ νομίζω πως η απάντηση είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να αναγνωρίσουμε τον ρόλο που παίξαμε μέχρι τώρα. Και Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επί ίσης ώρες στη διαπραγμάτευση με το Αζερβαϊτζάν ως ε, εταίρη, αλλά δεν, θα μπορούμε, δεν μπορούμε εμείς να τους κάνουμε κήρυγμα. Το Αζερβαϊτζάν είναι στο κάτω-κάτω της γραφής κυρίαρχο κράτος. Θα έλεγα ωστόσο ότι δεν έχουμε κοινέ αξίε. Υπάρχει εκεί έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν. Να πω λοιπόν για την Κομισιόν ότι το Κοινοβούλιο για την ώρα ούτε εγκρίνει ούτε απορρίπτει αυτή την προτινόμενη συμφωνία σύνδεσης. Αλλά σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε γνώμη. Ευχαριστώ. Thank you very much, Chairman. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι γενικά συζητάμε την κατάσταση και τη σύγκρουση και θα ήθελα, όπως και στην προηγούμενη έκθεση να συγχαρώ την εισηγήτρια για την ισορροπημένη αυτή στάση που κρατάει. Αλλά για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σας πω ότι υπήρξε προόδο τα τελευταία 3-4 χρόνια. Είμαστε η ωραία κοιμωμένοι βέβαια στην ε, όλη περιφέρεια. Αλλά σιγά σιγά γινόμαστε λίγο πιο δραστήριοι. Δεν νομίζω ότι ότι στέκει. Καλό φυσικά είναι που συμμετέχει η Ρωσία και διοργανώνει η κρίση όλες αυτές τις ε, συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Τι κάνουμε εμείς όμως. Ε, γίνονται συναντήσεις χωρίς αποτελέσματα όμως. Και νομίζω ότι το είδαμε αυτό και στην ανακοίνωση της ε, Επιτροπής ότι θα πρέπει να υπάρξει πιο έντονη εκπροσώπηση σε τομείς όπου δεν υπάρχει ε, έντονη εκπροσώπηση ακόμη. Όπω για παράδειγμα στη σύγκρουση του Ναγκόρνου Φραμπάχ. Άρα, γιατί να κάνουμε πίσω. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την ε, ανάπτυξη εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υποβοηθήσουμε την εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων. Παράλληλα να είμαστε αντικειμενικοί, να μην δημιουργήσουμε την ε, αίσθηση ότι προτιμούμε τον έναν υπέρ του άλλου αλλά ότι είμαστε υπέρ του διεθνού δικαίου. Γιατί είναι προ το των δύο χωρών να λάβει ένα τέλο αυτή η σύγκρουση και υπέρ τη Ρωσία μακροπρόθεσμα. Αν και φυσικά βραχυπρόθεσμα υπάρχουν και άλλε σκοπιμότητε. Σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά project τώρα, είναι κρίσιμο. Με τον αγωγό Ναμπούκο ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί εργασίες. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ολοκληρωθούν, οι αγωγοί να ολοκληρωθούν για το προς των πολιτών μας. Κυρία Μακοβέ, ευχαριστώ. Η συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής του Αζερβαϊτζάν από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία του και την εθνική του κυριαρχία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει τη χώρα να αυξήσει την ευημερία των πολιτών, να αναπτύξει την οικονομία, να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση όσο και η δικαιοσύνη. Όπως γνωρίζουμε, το Ζερμπαντζάν ε, είναι χώρα που αναπτύσσεται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στην οικονομία. Ε, Παγκοσμίω, όχι μόνο στην περιοχή. Από το 2004 ε, βλέπουμε αύξηση 300% παντού, όχι μόνο στο πετρέλαιο. Και επίσης διαφοροποιεί και τους τρόπους και τις οδούς παροχής ενέργειας προς την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, Υπάρχουν προκλήσεις σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και αλλού θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά θέματα, παραμένουν ακόμα και απομένουν πολλά να γίνουν για να βελτιωθεί ο τρόπος ε, πρόσληψης και διορισμού των δικαστών, ε, των εισαγγελέων με ε, ορθά κριτήρια και αντικειμενικά. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει ένα μητρό διώξεων και καταδικών για να μπορέσει ο καθένας να διαπιστώσει την πρόοδο για να βελτιωθεί και η δημόσια εμπιστοσύνη. Περιπτώσεις υψηλού επίπεδου διαφθοράς θα πρέπει ε, να ε, κρίνονται στα δικαστήρια. Και βεβαίως χωράει και πολύ βελτίωση η διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και στις δημόσιες δαπάνες η καταπολέμηση της διαφθοράς και οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντικές και να σας πω γιατί. Μετά από την εμπειρία αυτή των τελευταίων 20 ετών είναι εύκολο, πιο εύκολο να φτάσει κανείς στην οικονομία της αγοράς και σε άλλα στοιχεία της αγοράς. Είναι πιο εύκολο από το να γίνουν οι δικαστικές μεταρρυθμίσεις που φαίνεται ε, ότι είναι οι δυσκολότερες. Σε διεθνές επίπεδο το Αζερμπαϊτζάν είναι μέλος ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας, όχι μόνιμο, στον ΟΗΕ για το 12 και το 13. Ελπίζω αυτό να συνεισφέρει θετικά για τη διατήρηση της ε, ειρήνης και της ασφάλειας. Ε, το Ναγκόρνο Καραμπάχ παραμένει σοβαρό εμπόδιο για την ειρήνη και την ευημερία στην περιφέρεια του Νοτιού Καυκάσου και είναι και πρόκληση και για την ασφάλεια και για τη σταθερότητα σε όλη την Ευρώπη. Χρειάζεται επιγόντως επίλυση και ειρηνική διευθέτηση ε, της σύγκρουσης. Θα πρέπει να γίνει αυτό με βάση τις αρχές και τους νόμους του διεθνούς δικαίου. Και είμαι υπέρ των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι για να επιτύχουν αυτά θα πρέπει όλες οι πλευρές να ε, δείχνουν καλή πίστη και να σέβονται τις δεσμεύσεις και ε, τις υποσχέσεις τους και να τηρούν και τα σύμβεφονηθέν. Ευχαριστώ. Κυρία Λούνατσακ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Γέτερ Μάκη για το σχέδιο έκθεσης και για τα όσα μας παρουσίασε τώρα μόλις. Ε, μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας, μεγάλα έσοδα και λόγω του πετρελαίου και του φυσικού αερίου το Αζερβαϊτζάν ε, εμφανίζεται πλέον ως ισχυρός οικονομικός παράγων στην περιοχή αλλά ε, βλέπουμε και τις ελλείψεις που υπάρχουν στη δημοκρατία. Είναι πολύ σημαντικά και αυτά είναι τα ξέρετε. Δεν θα πρέπει να προωθείτε μόνο το ένα και να αγνοείτε, να παραγνωρίζετε το άλλο. Έχω την ε, αίσθηση ότι στον Ταβός ε, τους επενούν πάρα πολύ για τα οικονομικά τους επιτεύγματα και λιγότερο για τα υπόλοιπα. Για το θέμα της συμφωνίας σύνδεσης με το Σερβαϊτζάν, επιτρέψτε μου να κάνω μερικά σχόλια. Έχω την εντύπωση ότι σε αντίθεση με την Αρμενία, η αζερική κυβέρνηση δεν ε, διαπραγματεύεται με την ίδια ένταση ούτε δείχνει πάντα την ίδια προθυμία και τη βούληση να κάνουν πάρα πολλά. Δηλαδή του στυλ οικονομικά δεν χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε αρκετά έσοδα. Οπότε δεν έχει μεγάλη σημασία για μας να προχωρήσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι λέγουν Ας συνεχίσουμε ε, τη Συμφωνία Εμπορικής Συνεργασίας ε, και εταιρική σχέση δεν ενδιαφέρονται να αλλάξουν η μορφή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον αυτή η αίσθηση δημιουργείται. Και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε και να διαπιστώσουμε ότι είναι ένα παράγων ο οποίο επίση ε, ισχύει και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στι σκέψει μα κατά τη διαπραγμάτευση. Έρχομαι στα επιμέρου σημεία, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν για την Αρμενία. Πάρα πολύ σύντομα, αντίστοιχα ισχύουν και εδώ. αφού η χώρα είναι μέλος στην Ανατολική Γειτονία και γενικά από πλευράς Κοινοβουλίου θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν και σε αφοπλισμό αλλά και να γίνουν πρόοδοι στις διαπραγματεύσεις για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και να τα λέμε ειλικρινά αυτά τα πράγματα και με σαφήνεια. Γιατί σε τελική ανάλυση έχουμε μια εταιρική σχέση μαζί τους και βλέπουμε και τις συγκρούσεις ποιες είναι. Έχει νόημα το κοινοβούλιο ε, να τα λέει αυτά με στεναρό τρόπο. Ε, ε, σας επισημάνω και μερικά άλλα στοιχεία όπως τελευταίες εκλογές το 2010 ο ΑΣΕ προχώρησε σε μια σειρά συστάσεων για το τι πρέπει να βελτιωθεί στο μέλλον και σε αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε, να υλοποιηθούν τα συμπεράσματα και συστάσεις του ΑΣΕ. Κάποια άλλα θέματα τα οποία τα έχουμε σημειώσει και σε άλλα κείμενα για το Σερβαϊτζά και δεν συμφωνούσαν ε, οπωσδήποτε πάντα όλες οι πολιτικές ομάδες, αλλά εγώ θέλω να τα πω. Ο ειδικό εντεταλμένος ε, της κοινοβουλευτικής συνέλευσης ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους πολιτικούς κρατουμένους δεν επιτρέπεται, δεν του επιτρέπεται είσοδο στη χώρα. Εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή να μεταβεί γιατί υπάρχουν ε, κρατούμενοι στις φυλακές που κατά την άποψή μου είναι πολιτικοί κρατούμενοι και καλό θα ήταν να το θέτουμε και αυτό υπόψη τους. Ενδεχομένω, βέβαια αυτό δεν αναφορά την έκθεση, ε, αλλά να σκεφτούμε μήπως... μη γελάσετε σας παρακαλώ να ε, ε, ε, μπλοκάρουμε τη Eurovision που θα γίνει στο Αζερβαϊτζάν. Ξέρετε ότι κέρδισαν πέρσι, θα μπορούσαμε και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό για θέματα ανοίγματο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να τους απειλήσουμε ότι δεν θα γίνει Eurovision στον Πακού, γιατί θέλουν να προβάλλονται ως σύγχρονη χώρα, ε, ανοιχτή, γιατί όχι, να το σκεφτούμε. Δεν λέω να γίνει οπωσδήποτε τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή. Ανθρώπινα δικαιώματα, αφοπλισμός, τα είπα αυτά. Κάτι που με ενδιαφέρει και με απασχολεί και μένα είναι το εξή. Θα ήταν ε, χρήσιμο και σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει ε, προγράμματα και στις επίμαχες περιοχές. Ξέρω ότι η κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν το θεωρεί αυτό αναγνώριση ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης των εδαφών, αλλά για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό αυτό θα είχε νόημα. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω και για την Αρμενία και για το Αζερβαϊτζάν είναι η σύμβαση για, κατά των αρκών κατά προσωπικού. Θα πρέπει να προσυπογράψουν. Νομίζω ε, καλό θα ήταν και για τις δύο χώρες και θα είχαν συμφέρον να το πράξουν. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα ναρκοπέδια. Αυτά τα λίγα θα γίνει και δεύτερη συζήτηση. Μάλιστα. Καλά κάνατε και σταματήστε γιατί έχουμε πολύ σημαντικό θέμα που ακολουθεί και ε, συγητή και γνωμοδότηση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, να είμαστε πάρα πολύ σύντομα. Όταν θα έρθουν οι τροπολογίε θα τα ξαναπούμε και όταν οι εισηγητέ θα έχουν μεταβεί στην περιφέρεια εκεί, θα έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. η Κοίταξια. Τα άλλα, τα άλλα. Ναι, εδώ κάθομαι, κύριε Μπρόκο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρατηρήσεις σας. Για τις θέσεις που μας παρουσιάσατε. Αναμένω τις τροπολογίες σας και θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το κείμενο όσο πιο ισορροπημένο γίνεται. Και προσβλέπω λοιπόν στις ε, τροπολογίες που θα λάβω. Μάλιστα, ο πρόεδρος. Ξέρω ότι πάντα η Γυναίκε είναι πιο συνοπτικέ και σύντομε από ότι άντρε, αλλά πραγματικά ήταν υποδειγματική η κυρία Γιατεμάκη. Να παρακαλέσω όλους όσοι δεν ε, έχουν δικαίωμα συμμετοχή να εξέλθουν τις αιθούσε, γιατί η συζήτηση θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Μικρή διακοπή.